Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ε, ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου γύρου ψηφοφοριών. Λοιπόν, τα αποτελέσματα του τρίτου κομματιού του ψηφίσματος για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πανδημίας είναι τα εξής. Τροπολογία 42. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Δεκτή. 21. Απορρίπτεται. 69 απορρίπτεται 70 απορρίπτεται 47 δεκτή 4 δεκτή 71 απορρίπτεται 12 απορρίπτεται 5 δεκτή 26 δεκτή 72 απορρίπτεται 27 δεκτή 6 δεκτή 73 απορρίπτεται 23 δεκτή 74 Δεκτή. 75. Απορρίπτεται. 79. Απορρίπτεται. 714 και 27 ταυτόσημες δεκτές 20 δεκτή παράγραφος 36 3 μέρη μέρος πρώτο δεκτό Δεύτερο μέρος. Δεκτό. Τρίτο μέρος. Δεκτό. 37. Αρχικό κείμενο. Μέρος πρώτο. Δεκτό. Μέρος δεύτερο. Επίσης δεκτό. 50. Δεκτή. 16. 51 απορρίπτεται και τέλος 52 επίσης απορρίπτεται τα αποτελέσματα της τέταρτης ψηφοφορίας για το κοινοψήφισμα για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πανδημία και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν αύριο το πρωί στις 9 όταν θα επαναληφθεί δηλαδή η συνεδρίαση. Έχει δημοσιευτεί η ημερήσια διάταξη στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λύεται εδώ η συνεδρίαση. Καλή ξεκή, ξεκούραση σε όλους και ευχαριστώ τις υπηρεσίες που δουλεύουν τόσο αργά. Λύεται η συνεδρίαση.